Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θα αρχίσουμε τη ε, συζήτησή μας με την παρέμβαση του κυρίου Ρόελ, ο οποίος είναι συντάκτης της προφορικής ερώτησης. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε για πέντε λεπτά. Herzlichen Dank, guten Morgen